Bien, mes chers collègues, nous reprenons αγαπητοί συνάδελφοι. Και σήμερα, λοιπόν, στην ημερήσια διάταξη έχουμε καταρχά ε, το θέμα τη ενημέρωση από πλευρά του εισηγητή μα για τον Γενικό Προπολογισμό του 2017 για όλα τα τμήματα. Θα γίνει λοιπόν ε, η συζήτηση και στι 10.30 θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τι εργασίε μα. Δεν έχω ανακοινώσει να σα κάνω. Και αν είναι έτοιμο ο κύριο Γκάιερ, α πάρει πάρα αυτό το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σας έχω καταρτήσει και ένα έγγραφο, το οποίο νομίζω το έλαβαν και οι σκιώδεις και οι συντονιστές. Πρόκειται για την πρόταση την δική μου για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις 2.200 ε, τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από τις επιτροπές, από τους εισηγητές, αλλά και από πολλούς μεμονωμένους βουλευτές. Το έγγραφο λοιπόν αυτό από χτε ήδη είναι ξεπερασμένο ενδεχομένω, πρέπει να σας πω. Γιατί ξέρετε, πολιτικός και πραγματικός, πώς να σα το πω, ήταν δύσκολο να ολοκληρώσουμε αυτές τις εργασίε τις οποίες μας ανέθεσε η κυρία Γεωργίευα χθε ε, και θεωρώ ότι σε γενικέ γραμμέ είχαμε σημειώσει γενικώ πρόοδο. Και φυσικά έχει σχέση ιδιαίτερα αυτό με το έγγραφο που έχω κατατήσει. Αλλά δεν αποτυπώνονται αυτά τα οποία οι πιο πρόσφατες εξέλιξεις στο έγγραφο αυτό. Να ευχαριστήσω καταρχάς ε, τους συναδέλφους από τη γραμματεία της Επιτροπής γιατί το Σάββατο και οι δύο πλευρές ε, θυσίασαν το μισό του Σαββατοκύριακο για να καταρτήσουν ε, τη βάση, τα θεμέλια του εγγράφου αυτού και εξετάσαμε επισταμένως τις τροπολογίες, κοιτάξαμε το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε, το τι θα έβγαζε νόημα πολιτικά, από πολιτικής άποψης. Και αυτό ασφαλώς ήταν πολύ χρήσιμο. Γιατί χωρίς αυτή την ε, φάση θα ήμουν χαμένος ε, ως ε, εισηγητής για τον προϋπολογισμό και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους που ε, εργάστηκαν σκληρά για την προετοιμασία του εγγράφου αυτού για να γίνει και το debriefing. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά τους. Δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από πλευράς μου και προς τους βοηθούς μου που δεν είναι εδώ, αλλά και προς ε, τις συναδέλφους μου, γιατί κυρίως γυναίκες είναι, πρέπει να σας πω, από πλευρά των σοσιαλιστών, οι οποίοι πραγματικά με βοήθησαν εντυτέρως. Σας είπα λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως πρέπει να τα εξετάσουμε εκ νέου μετά από, από αυτά που μας παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άρα είναι ενδιαφέρουσα η πρόκληση και από πολιτική άποψη και από διανοτική άποψη, αν θέλετε. Τα κομμάτια του πακέτου τα οποία μα παρουσίασε χθε η κυρία Γεωργίεβα, τα οποία τα υποστηρίζουμε, θα πρέπει του επόμενου μήνε όχι μόνο να τα περάσουμε, αλλά. Θα επανέλθω και σε κάποια σημεία. Γιατί ενδεχομένω στην αναθεώρηση του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαίσιου να έχουν επηρεάσει κάποια στοιχεία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να εναρμονιστούν. Αυτό θα είναι δύσκολο και από τεχνική πλευρά, αλλά και πόσο μάλλον που θα υπάρχουν και πολιτικέ ε, αλληλεπιδράσει. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά θα αποτελέσει ε, μια επιπλέον δυσκολία. Θα δούμε και τι θα προκύψει από την αματεργασία του κ. Μόντι σίγουρα θα προσθεθούν και από εκεί σημαντικές λεπτομέρειες. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά. Τώρα, πολλά στοιχεία τα γνωρίζετε και από τις προηγούμενες διαδικασίες για την προπολογισμό. Και εγώ πιστεύω ότι όλες οι γραμμές του προϋπολογισμού που τροποποιήθηκαν από το Συμβούλιο θα πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι άλλο που το ξέρουμε και από το παρελθόν, επίσης, είναι η, πρόσταση, η πρόταση για τα εφιστάμενα μέσα, contingency, margin, συνολικό περιθώριο για τις δεσμεύσεις, να κινητοποιηθούν για να ενισχύσουν κάποιες ε, αμφιταραντευόμενες και κρίσιμες ε, γραμμές του προπολογισμού. Σε ό,τι αφορά το ΣΕΦ και την, ε, τον ορίζοντα 2020 προτάθηκαν περικοπές. Αυτό στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να ανατραπεί, να, συνα, ε, να συνεχιστεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και πολλές καλές ιδέες που περιλαμβάνονται στα, στα προγράμματα να περάσουν. Και αυτό με οδηγεί στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι λίγο αμφιλεγόμενο και λίγο προκαλεί διάσταση απόψεων και στη δική μας Επιτροπή. Θέλω να σας το παρουσιάσω σαν δική μου τοποθέτηση. Δεν είναι φυσικά κανόνας απαράβατος ε, στην παρούσα φάση, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλούσω να σας παραθέσω την επιχειρηματολογία μου για το θέμα αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει μία πρόταση για ένα μέτρο ε, προετοιμασίας για την κινητοποίηση 30 δισεκατομμύριων ευρώ ε, επί τρία έτη για την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Εξοπλισμών. Πρόκειται για ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο μιας ε, αναπτυσσόμενης κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας που θα συζητηθεί και στην Πρατισλάβα σήμερα αύριο. Δεν είναι τυχαίο ω στοιχείο, δηλαδή πρόκειται για μια εφαρμογή μιας ιδέας Δεν πρόκειται για μια τυχαία ιδέα, μάλλον ενός τυχαίου δημιουργού. Όχι, πρόκειται για ένα ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας. Και αυτό πολιτικός πώς θα μας περάσει στο επόμενο επίπεδο, θεωρούμε. Προσωπικά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση δεν περνάει και την καλύτερη φάση της και άρα ενδεχομένως να μην χρειάζεται μια κοινή πολιτική ασφάλειας και μια πολιτική άμυνας για να ανακάμψει. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό και άρα θα πρέπει να προστατευτούμε από, τους εξωτερικούς, από τις εξωτερικές απειλές. Αυτό στέκει. Άρα δεν έχω επί του περιεχομένου οποιαδήποτε αντίρρηση. Εκεί που έχω προβλήματα είναι στο θέμα της χρηματοδότησης. Θα πρέπει απλά να έχουμε υπόψη μας το εξή. Τα 90 εκατομμύρια στον επόμενο προπολογισμό και υπάρχει υποχρέωση 25 από αυτά τα 90 εκατομμύρια θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, μάλλον θα σήμερα ότι δεν θα μπορεί να χρηματοδοτηθούν σημαντικά πολιτικά προγράμματα και σημαντικές ε, άλλα προγράμματα, άρα πολιτικά. Θα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση. Καλούμαστε πολιτικά να λάβουμε απόφαση για το ποια πιλωτικά προγράμματα και τι προπαρασκευαστικές δράσεις αξίζουν να ενισχυθούν και αν τα προπαρασκευαστικά μέτρα για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι από αυτά τα μέτρα, αυτόματα το ποσό που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα είναι χαμηλότερο. Αυτό είναι αυτοματισμός. Και στην παρούσα φάση λοιπόν έχω να κάνω μία πρόταση. Μία πρόταση η οποία προκύπτει, αν θέλετε, και πηγάζει από την εξή ιδέα. Γνωρίζετε ποια είναι η στάση μου, την έχω παρουσιάσει πολλά και εδώ στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Πιστεύω ότι... Κοιτάξτε, έγινα Ευρωπαίος πολιτικός γιατί πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορεί να κάνει η πολιτική και συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους με τη συνεργασία τους για να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό αποτυπώνεται στον προπολογισμό, αλλά δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο αυτό ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται. Έχουμε πάρα πολλά κοινά καθήκοντα τα οποία πρέπει να εκτελέσουμε και τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία μας διαθέτουν τα κράτη-μέλη, από τα οποία και εξαρτώμαστε άλλωστε, πολύ απλά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Αυτό ενδεχομένω να βελτιωθεί μετά τη χθεσινή πρόταση, όπω την ακούσαμε, αλλά Το κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτό και στον προπολογισμό είναι κάτι το αμφιλεγόμενο. Δεν έχει γίνει έως τώρα. Και νομίζω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση ξεκινούμε. Υπάρχουν ε, και άλλοι μηχανισμοί, μηχανισμός ε, των Αθηνών για τη χρηματοδότηση της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχουν αυτά τα μέσα, Αν αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό τα μέσα για την κοινή πολιτική ασφάλεια και την πολιτική άμυνα, παρά το γεγονό ότι θα έχει νόημα αυτό, θα ανοίξουμε του ασκού του αιώλου. Και θα έρχεται διαρκώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα παρουσιάζει πολιτικώ ορθέ προτάσει και εμεί πολιτικά θα μα λένε, κοιτάξτε, μια και βγάζουν νόημα όλα αυτά τα μέτρα, να τα υποστηρίξετε. Αλλά η πραγματικότητα από πλευρά προπολογισμού και χρηματοδότηση είναι ότι ε, μάλλον δεν θα έχουμε τα ποσά αυτά. Και ανεξάρτητα από αυτά που μας είπε η κυρία Γεωργίεβα χθες, εγώ πιστεύω ότι δεν τα έχουμε τα μέσα αυτά. Δεν έχουμε τις, ε, τα χρήματα αυτά. Και άρα είμαι πολύ διστακτικός για τα μέτρα αυτά, τα προπαρασκευαστικά και την χρηματοδότησή τους. Από τους, ε, τον προπολογισμό. Κοιτάξτε, το λόμπι που μου ασκούν είναι αμήλικτο από την ε, γαλλική κυβέρνηση μέχρι την κυρία Χολμαϊρ και δεν ξέρω ειλικρινά ποιο είναι και πιο αποτελεσματικό από του δύο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έω τώρα αναζητώ άλλε χρηματοδοτικέ πηγέ και έχω και μία ιδέα να σα την παρουσιάσω να δημιουργηθούν αυτέ οι γραμμέ για τι προπασκευαστικέ δράσει, προκειμένου να δείξουμε ότι επί του περιεχομένου υποστηρίζουμε το έργο αυτό ή ιδάλλως θα μπορούσαμε απλά να το απορρίψουμε άρα να δημιουργηθεί αυτή η γραμμή του προπολογισμού και έτσι να υποστηρίξουμε ε, επί του περιεχομένου, επί τη αρχή το project αυτό, αλλά να βάλουμε μηδενικού πόρου, μηδενική χρηματοδότηση και να γράψουμε στη γραμμή του προπολογισμού αυτή ότι θα θέλαμε και έχουμε λίγο χρόνο για να έχουμε κάποιες ε, άλλες ε, ε, προτάσεις για τη χρηματοδότηση. Μπορούμε να προτείνουμε το μηχανισμό των Αθηνών, τις εξωτερικές, τα εξωτερικά έσοδα, τεχνικές αλλαγές. Αλλά να δώσουμε καταρχάς το μήνυμα ότι θέλουμε και υποστηρίζουμε αυτό το project και κατά δεύτερο να δώσουμε το μήνυμα ότι ο προϋπολογισμός αυτός πολύ απλά δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοια μέτρα και κατά τρίτον ότι αν τα κράτη-μέλη επιθυμούν να υπάρχουν αυτή κοινή, αυτό το κοινό εγχείρημα θα πρέπει να συμμετέχουν ε, στη χρηματοδότηση. και θεωρώ ότι αυτό θα είχε καθοριστική επίδραση στο Κοινοβουλίο γιατί θα μας ε, έβαζε σε θέση να χρηματοδοτούμε πιο πολλά πλαιτικά προγράμματα και πιλωτικέ δράσεις. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα σε ό,τι αφορά το τμήμα 1α το οποίο επηρεάζεται από όλα αυτά που σας περιέγραφα μέχρι τώρα. Έχουμε την εξή πρόταση. Οι γραμμές του προπολογισμού να τις επαναφέρουμε στο επίπεδο πριν του ΕΦΣΙ σε ό,τι αφορά τον ΡΙΖΟΝΤΑ 2020 και το Connecting Europe Facility και Θα ήθελα και στο τέλος να πω και κάτι για την κατηγορία 1α ή το τμήμα 1α, αλλά 50% των κονδυλίων για το 2017 για το ΕΦΣΥ θα πρότεινα να μπουν στο αποθηματικό. Γιατί σε ό,τι αφορά το Εράσμου στο κόσμο και το ΟΗΡΕΣ, ε, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να γίνει η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες που έχει η ΕΝΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την ε, ασφάλεια δικτύων, να βελτιωθούν αυτές οι δυνατότητες. Για να ανταποκριθούμε σε όσα ζήτησε η ΕΚΟΝ. Η δημιουργία παθηματικού σε ό,τι αφορά ε, αυτά που προέκυψαν και από τους οικονομικούς ελέγχους και να δημιουργηθεί μια γραμμή προϋπολογισμού για ειδικά, ειδικές εκδηλώσεις. Γιατί? Γιατί πολλοί συνάδελφοι, κυρίως Αυστριακοί, που θα γίνουν οι επόμενοι παραολυμπιακοί, ζητούν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ζητήσουν ευρωπαϊκούς πόρους. Εγώ θεωρώ ότι και δυνατό είναι αυτό και ευκταίο. Η λογική πηγή χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, δηλαδή του αθλητισμού στο εσωτερικό του Εράσμου, διατίθεται μεν, αλλά θα ήθελα να μας διαβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ενδεχόμενο αίτημα από πλευράς της Αυστρίας θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί επαρκώς. Άρα, δημιουργώντας αυτή τη γραμμή του προπολογισμού, ουσιαστικά εξασφαλίζουμε την χρηματοδότηση των ε, παραλυμπιακών. Θα ήθελα να λειτουργούσε αυτό από το Εράσμους και το κομμάτι που προορίζεται για τον αθλητισμό. Αλλά συμφωνώ και με τις αμφιβολίες που εκφράστηκαν. Μία γραμμή του προπολογισμού η οποία έχει σηματοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό ε, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για την κατεύθυνση αυτή, αλλά έχω πρώτο πρόβλημα. Αν ε, εμεί τελικά εφησυχαστούμε και υποθέσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί το Erasmus Plus και το κομμάτι για τον εθνικισμό και τελικά δεν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, να μην έχουμε θέματα με τη χρηματοδότηση των Παραλυμπιακών. Άρα θα κάνω διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δω τι δυνατότητες υπάρχουν για τη χρηματοδότηση από το Erasmus ε, Sport, από το κομμάτι του αθλητισμού δηλαδή του Erasmus αν μας διαβεβαιώσουν ότι είναι δυνατόν, μπορούμε να, να μην δημιουργήσουμε αυτή τη γραμμή προπολογισμού, αλλά ως εξασφάλιση το έχω σκεφτεί. Να αναφέρω ένα δεύτερο στοιχείο τώρα, το οποίο επικρίνεται ιδιαίτερως. Σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΙ συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του κ. Γιούγκερ. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θέλω να ζημιώσω το εργαλείο αυτό, το μέσο αυτό. Αυτό θα ήταν παράλογο. Κανείς δεν το ισχυρίζεται άλλωστε. Κανεί δεν θέλει να το βλάψει, γιατί η δημιουργία του ταμείου αυτού ήταν ε, και η προϋπόθεση που είχε θέσει η ομάδα μου για την εκλογή του Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργεί ωστόσο έτσι όπως θα το επιθυμούσαν όλοι. Δεν είναι ιδανικό. Και υπήρχε και μια πρόταση από την, από την Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων. Δεν είναι αυτό διαπίστωση μόνο τη ομάδα μου. Έχουμε το θέμα τη προστατικότητα. Ω τώρα λοιπόν, κοιτώντα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί το ΕΦΣΕ, βλέπουμε για παράδειγμα αυτοκινητόδρομου στη Γερμανία ω project. Είναι η Γερμανία η πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη. Περιφανεύονται οι πρωθυπουργοί μας ε, ότι δεν έχουμε υπερβολικό έλλειμμα. Αυτό λοιπόν ήταν αυτό που περιμέναμε από το ΕΦΣΥ. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με μια ισορροπία. Ένα πρόβλημα το οποίο το διέκρινα εξ αρχής και το οποίο ουσιαστικά τα κράτη-μέλη δεν το αναγνωρίζουν στην πλήρη του έκταση. Κοιτάξτε, είναι προφανές αγαπητοί συνάδελφοι οικονομικά ισχυρές χώρες με αναπτυσσόμενο οικονομικό κλάδο, αυτές οι χώρες επωφελούνται πιο πολύ από ένα μέσο, ένα ταμείο όπως το ΕΦΣΥ. Άρα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ αναπτυγμένες πρωτεύουσε που δεν τα πηγαίνουν τόσο καλά. Υπάρχουν, για παράδειγμα, ε, χώρες όπως η Γερμανία, όπου υπάρχουν ταμεία ενίσχυσης και υπάρχουν και χώρες που δεν έχουν ταμεία ενίσχυσης όπως η Γερμανία. Δεν μπορούμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντισταθμίσουμε τις διαφορές αυτές. σύμφωνα, αλλά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αυτό αυτή η έλλειψη ισορροπίας προκειμένου να ε, καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσπαθήσει κάπως να διορθώσει αυτή την ανισορροπία, βελτιώνοντας την τεχνική αρρωγή, την χρηματοδότηση σε χώρες που δεν έχουν τέτοιες ε, τράπεζες ενίσχυσης και το καθεξής. Και λοιπόν, ως βουλευτές θα πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Θέλουμε να τα παρουσιάσουμε αυτά στην ΕΤΕΠ και να ελπίσουμε να τα καταλάβει και να ελπίσουμε να τα εφαρμόσει ή θέλουμε το τελευταίο κοινοβουλευτικό μέσο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας να το χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση στην ΕΤΕΠ. Αυτό είναι το ερώτημα που έχω να θέσω. Και η απάντηση είναι η εξή. Σε ό,τι αφορά μέσα όπως το ΕΦΣΙ, δεν έχουμε κανένα κοινοβουλευτικό έλεγχο, καμία κοινοβουλευτική επιρροή. Και να σας πω ότι αυτό το α, μέσο Θέλουμε να συνεχιστεί. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα τα οποία από τη δομή τους, από τη σύνθεσή τους δεν επιτρέπουν κοινοβουλευτική επιρροή. Δηλαδή, στην αρχή έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε κάποιους όρους, κάποιες προϋποθέσεις, να πούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Στην αρχή μπορούμε κάπως να διαμορφώσουμε τα μέσα αυτά και έχουμε μισό έτος, ε, μισό χρόνο προσπαθούσαμε ως κοινοβούλιο κάπως να διαμορφώσουμε και εμείς το ΕΦΣΙ. Κάπως το βελτιώσαμε, δεν λέω. Αλλά τώρα που έχει ξεκινήσει και λειτουργεί πλέον το μέσο, δεν έχουμε κανένα περιθώριο να ασκήσουμε οποιαδήποτε επιρροή πέρα με κάποια επιχειρήματα. Αλλά κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, εφή επιχειρήματα έχουμε χρησιμοποιήσει σε πολλές περιστάσεις έναντι του Συμβουλίου και ξέρουμε τι θα κάνει το Συμβούλιο. Μπορεί να συζητάμε και να μου πείτε ε, σήμερα ότι «Α, κύριε Γκάιερ, λάθος κάνετε». Μια χαρά τα πάει το ΕΦΣΙ, φοβερό εργαλείο. Και έχουμε και επιρροή και μπορούμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο και να αποφασίσουμε τι θα γίνει. Εντάξει, κοιτάξτε, αν αυτή είναι η άποψη της πλειοψηφία, εγώ ε, θα το δεχτώ. Αλλά εγώ θα πρότεινα, αν θέλουμε να βελτιώσουμε το ΕΦΣΙ, Τώρα είναι η ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Και αν δεν την αδράξουμε, εντάξει. Ας το πάρουμε απόφαση, αλλά πιστεύω ότι ήταν πολιτικό λάθος. Κατηγορία 2 τώρα. Α, συγγνώμη. Τώρα σε ό,τι αφορά το τμημα ένα 1β πρώτα. πρόταση λοιπόν είναι η εξή. Στο τμήμα 1β και μάλιστα αυτό θα είναι το πιο σημαντικό που θέλω να σα αναφέρω σήμερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τομέα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Απασχόλησης. Ε, χρήση επιπλέον πόρων 1,5 δις. Και το ακούσαμε αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλαμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Αυτό είναι το βασικό το οποίο ε, πρότεινα. Δεν ήμουν ικανοποιημένο με το γεγονός ότι είχαμε προτείνει επιπρόσθετες πληρωμές και επιπρόσθετα μέτρα για να εξισορροπηθούν άλλες χρηματοδοτήσεις, αλλά πιστεύω ότι μετά την πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαπιστωθεί ότι το μέσο αυτό για την απασχόληση ε, θα τσουλήσει από μόνο του μετά τις πρώτες ε, δυσκολίες. Και γι' αυτό λοιπόν ε, συμφωνώ σε ό,τι αφορά τις ε, δεσμεύσεις. Τώρα, στο τμήμα, το δεύτερο, δεύτερο τμήμα. Και εδώ θέλουμε φυσικά να επανέλθουμε στα επίπεδα του σχεδίου προπολογισμού όπω προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τα όσα θεωρούνται απαραίτητα για τη χρηματοδότηση του πακέτου για την υποστήριξη έκρητης ανάγκης, ιδιαίτερα για τον γαλακτοκομικό κλάδο. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται και με τα ποσά τα οποία θα αφιερώνουμε στις γραμμές. Περιμένουμε το Νοέμβριο να δούμε και την διορθωτική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ξέρουμε ότι αυτό θα προσθέσει χρήματα στο τμήμα 2 και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Αυτά τα επίσης μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον αγροτικό κλάδο. Τώρα, αν αυτό το ποσό είναι μικρότερα από τα 500 εκατομμύρια που πρότειναν οι χριστιανοδημοκράτες. Θα πρότεινα να προσθέσουμε το ποσό που υπολείπεται. Συμφωνούμε απόλυτα και ομόφωνα στο ότι υπάρχει ανάγκη και στο ότι πρέπει να δράσουμε, αλλά το μόνο που με βρίσκει κάπως αντίθετο για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα 500 εκατομμύρια που ζητούν οι χριστιανοδημοκράτες ασφαλώς αποτελούν ένα μήνυμα σαφές. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά νομίζω ότι στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να βάλουμε ακριβή ποσά σε αυτή, τη γραμμή, γιατί θα λάβουμε και χρήματα από την ε, διορθωτική επιστολή και θα δούμε τι θα πρέπει να προσθέσουμε εκ των υστέρων μετά. Μάλιστα. Τώρα το τμήμα 3. Χαρακτηρίζεται όλος ιδιαίτερος το τρίτο τμήμα αυτό από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αξιοποιεί πλήρως τα περιθώρια για τη χρηματοπότηση όλων των μέτρων που θα χρειάζονταν στο πακέτο ασφαλείας. Το Συμβούλιο αρκετά μονόμερος έκανε επίθεση κατά των πολιτισμικών προγραμμάτων, έκανε περικοπές και νομίζω έβαλε ε, ένα συμβολικό αποθεματικό 27 εκατομμύρια. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω να το απορρίψουμε, να απορρίψουμε αυτή την πρόταση του Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγγνώμη, και να επανέλθουμε στα πέρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα πολιτισμικά προγράμματα είναι και προγράμματα συμβολικά, ξέρετε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν επιπλέον. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ευελιξία του πολιτισμού δημοσιονομικού πλαισίου προτείνω να υποστηρίξουμε την ε, Europol και την ΕΑΖΟ και επίσης ευρωπαϊκό έτος κοινή πολιτισμικής κληρονομιάς ελπίζω να υποστηριχθεί αυτό το πρόγραμμα και για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης. Αυτό δεν χρήζει ξεχωριστής ε, οικονομικής ενίσχυσης, ε, μπορεί να ενταχθεί στο ESF και να χρησιμοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί από αυτό. Και ένας ε, ευρωπαϊκός μηχανισμός για την υποδοχή των προσφύγων που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το ΆΜΕΦ σε ό,τι αφορά το τέταρτο θέμα. Και αυτό περίπλοκο ζήτημα. Από τον τίτλο τι βλέπω. Και τη διαπιστώνω ότι ανησυχώ, ανησυχώ το τι θα μείνει τελικά από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ανάπτυξη. Γιατί τα πιο βασικά μέσα τα οποία έχουμε για την άσκηση πολιτική ανάπτυξη μειώνονται. Η δεύτερη δόση, για παράδειγμα, για τη χρηματοδότηση τη δεύτερη δόση του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες. Γιατί σκοπός μας είναι να διαθέσουμε κονδύλια προς την κατεύθυνση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το στοιχείο για την προταξική βοήθεια ε, και την πολιτική γειτονία να επηρεαστούν αυτά. Και σε τελική ανάλυση έχω να πω το εξή. Ε, ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα μέσα αυτά ε, δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να αυξηθούν εκ νέου οι πρικοδοτήσει των προγραμμάτων αυτών. Γι' αυτό τα προγράμματα τα οποία έχουν περικοπεί θεωρώ ότι θα πρέπει να επανέλθουν στα αρχικά επίπεδα που προβλέπονταν. Και η γραμμή του προπολογισμού. που ήταν στο παρελθόν προτεραιότητες να ενισχυθούν επίσης επιπρόσθετα σε ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη της τουρκικής κοινότητας στην Κύπρο γραμμές συγκεκριμένες ε, στο DCI αλλά και το όνρα, τη βοήθεια στους Παλαιστίνιους προσφύγους και τέτοια πράγματα. και από πλευράς της Επιτροπής Ανάπτυξης και από τους ε, φιλελεύθερους ε, μου ζητήθηκαν ε, νέες γραμμές προϋπολογισμού για την υποστήριξη των trust funds, των καταπιστευμάτων. Και θα είχα και άλλη μια πρόταση να κάνω. Στο τμήμα 4 αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τα ποιοτικά προγράμματα. Αυτό είναι τεχνική πρόταση, αλλά έχει και πολιτικές διαστάσεις. Υπάρχει, υπάρχουν οι ειδικοί αντιταλμένοι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δαπάνη των οποίων έω τώρα χρηματοδοτούνταν από την, το τέταρτο τμήμα. Αλλά αυτό ε, δεν είναι απαραίτητο, γιατί στην τελική ανάλυση ε, πρόκειται για προσωπικό το οποίο πληρώνεται από τη διοίκηση. Άρα θα πρότεινα αυτοί οι ειδικοί εντεταλμένοι να βγουν από το τέταρτο τμήμα και να μπουν στο πέμπτο τμήμα. Αυτό θα μας έδινε κάποια ευελιξία, κάπου 50 εκατομμύρια νομίζω, στην, ε, στο τέταρτο τμήμα. Συνάδελφοι, θα το ξέρεις καλύτερα από μένα αυτό το πόσο. Και αυτά τα μέσα που θα απελευθερώνονταν θα μας ε, επέτρεπαν στο τέταρτο τμήμα να τα βγάλουμε κάπως καλύτερα πέρα σε ό,τι φορά τα τα μέτρα. Στην πέμπτη, στο πέμπτο τμήμα τώρα. Αυτό είναι ε, αρμοδιότητα του συναδέλφου Τάραντ και άρα θα περιοριστώ στο να πω το εξή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επανέλθουμε και επανέλθαμε δηλαδή στην πρότασή μας στα επίπεδα της, ε, του σχεδίου προϋπολογισμού όπως τον πρώτον Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι έτσι ολοκλήρωσα τα όσα είχα να σας πω. Merci, monsieur le rapporteur général. Merci pour, euh, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα κάνατε εσείς και ε, οι συνεργάτες σας, ε, κυρίως ε, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πραγματικά πρώτη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι άθλος να είναι κανείς εισηγητής. Ο κύριος Στάρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αρχίζω με ο, κάπως εγωκεντρικά, δηλαδή θα ασχοληθώ με το ίδιο το κοινοβούλιο πρώτα απ' όλα. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία στις πολιτικές ομάδες ε, για δημιουργία 76 νέων θέσεων. Ε, πάντως είμαι, εγώ ανήκω μάλλον σε, σε μειοψηφία. Πρώτη φορά δε διαφωνούμε. Βλέπετε ότι για ζητήματα δημοσιονομικά είναι αρκετά συγκρουσιακό το κλίμα. Το Κοινοβούλιο αποκαθιστά πολλές γραμμές που περιέκοψε το Συμβούλιο και Κυρίως πρέπει να υπερασπιστούμε τα περί δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ενώ είχε ληφθεί απόφαση και από το Συμβούλιο τώρα περικόπτει τα κονδύλια για τις βασικές λειτουργίες του δικαστηρίου. Τώρα οι συνάδελφοι από την ΑΦΕΤ ε, ασχολήθηκαν με το προσωπικό στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η πρόταση για 16 ε, νέες θέσεις ε, στη Μονέα Μονάδα Στρατηγικής Επικοινωνίας, το υποστηρίζω, υποστηρίζω αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε ο Γκάιερ, ότι αν συμφωνεί, γιατί υπάρχει και πρόταση να μπει στο, ο ειδικό ε, απεσταλμένος στον προϋπολογισμό της ε, ε, δράσης. Α, ναι. Θα ήθελα την υποστήριξή σας ε, για να αποκατασταθεί η γραμμή για τον επόπτη, για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτά, Πρόεδρε. Merci, merci, monsieur. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Για τους ε, οργανισμούς. Monsieur Gaillard. Εκεί, τώρα, σε ό,τι αφορά τις, ε, αυτές τις ε, οργανισμούς της εξωτερικής υπηρεσίας. Αυτό έχει διαγραφεί στην πρώτη πρόταση. Αλλά ουσιαστικά τι προτείνω να ανατραπούν οι περικοπές που έκανε το Συμβουλίο και ως γενική γραμμή προτείνω όπου οι εξωτερικές υπηρεσίες έχουν ήδη ε, συνδράμει για την, ε, συμβάλει για την μείωση του προσωπικού κατά 5% να επανέλθουμε στα προγράμματα τα και στο, στις προβλέψεις που προβλέπονται στο 2016. Στο 1α προτείνω πιο πολλά χρήματα για την ΕΝΙΖΑ και στο τρίτο τμήμα για την Europol και την Eurojust και την ΕΑΖΟ προτείνω πιο πολλούς πόρους, πιο πολλά κονδύλια. Και σε ό,τι αφορά τα σχέδια ε, συστάσεις ε, στα πλαίσια Europol ε, γίνεται μια πολύ επικρατική συζήτηση σε ό,τι αφορά ε, αυτά που αποφάσισε η Επιτροπή για τις ελευθερίες του πολίτη και που θα ήθελε να έχει αποφασίσει. Υπάρχει μια σύγχυση. Δέκα θέσει στην ε, ε, Europol, δώδεκα στην... Έξι στην Ενίζα και δώδεκα στην Europol. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλα σημαντικά ζητήματα, θεωρώ ότι αρμόζει αυτή η αύξηση προσωπικού. Αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο για τις εξωτερικές υπηρεσίες. Ε, συγγνώμη, για τα, τώρα για τα ειδικά ε, μέσα, χρηματοδοτικά μέσα. Εδώ και τα ειδικά αυτά χρηματοδοτικά μέσα ε, η πρόταση είναι για το αποθεματικό κατά ανάγκη ανάγκης να αυξηθεί σε ένα δί Και προσδοκίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση. Θα πρέπει φυσικά να δούμε και τις χθεσινέ προτάσει τι ακριβώς περιλαμβάνουν. και το σχέδιο προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμίωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Και αυτό είναι επανέλθει στα επίπεδα του σχεδίου προϋπολογισμού. Και οι πληρωμέ. Και εκεί να ανατραπούν οι περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο, ως γενική αρχή οι δεσμεύσεις πληρωμών θα πρέπει να επαναληφθούν στα επίπεδα του σχεδίου προπολογισμού και στους τομείς εκείνους όπου έχουν αυξηθεί οι δεσμεύσεις ε, πληρωμών, εκεί τουλάχιστον που πιστεύουμε, κυρίως μάλλον που θεωρούμε, ότι οι πλήρωμες και οι προσδοκίε πληρωμών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απεσιόδοξε σε ό,τι αφορά και την χορήγηση των μέσων. να δημιουργηθεί μια, μια διαφορετική ισορροπία, να υπάρχει δηλαδή 100% δυστυχία μεταξύ των δεσμεύσεων και των πραγματικών πληρωμών. και με την ε, αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία γιατί η Επίτροπος ε, Γεωργίβα είπε ότι ενδεχομένω να δεχτεί τα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που είναι ε, υπέρ του ανωτάτου ορίου ακόμη και για τις πληρωμές. Ίσως το Συμβούλιο το ίδιο να προωθήσει αυτό το όραμα και να καθιερωθεί ήδη από το 2017. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Για να ακούσουμε τους κοιόδης τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, συνάδελφοι. Και από τις δικές μου πλευράς να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή για τη δουλειά του τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά επίσης και για το πόσο συνεργάσιμος ε, ήταν εμάς τους ε, σκιώδους με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Αυτό το οποίο θέλει ο ΛΟΑΣΕΛ ε, είναι αυτό το οποίο αποτυπώσαμε εσείς στον πολιτισμό στην ομάδα από τα πρώτα λέμε ότι το σχέδιο προπολογισμού που υπευλήθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη του Ιουνίου ήταν ένας ε, προϋπολογισμός λιτότητας αλλά είναι δεδομένες οι προτεραιότητές μας αυτές που είμαστε στην αρχή της περίοδου του MFF απασχόληση, ανάπτυξη, μεταναστευτικό και ασφάλεια για τους Ευρωπαίους. Οπότε θεωρούμε ότι το σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν πολύ πιο δόκιμο από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ως πολιτική ομάδα ότι δεν θέλουμε να δεχθεί το Κοινοβούλιο τίποτα από προτείνει το Συμβούλιο. Αυτό το είπε και ο πρόεδρος της ομάδας μας και το είπαμε και τις πρόσφατες εβδομάδες και είπαμε ότι από εκεί ξεκινούμε, είμαστε κατά αυτών των περικοπών του Συμβουλίου. Και συμφωνούμε με τον εισηγητή από αυτού. Κάτι άλλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, γι' αυτό καταπληκτούμε και τροπολογίες, έχουμε την έκθεση ε, για την αναθεώρηση του πολιτού πλαισίου. Άλμπριχ και το Μάνι συνέλφοι που κατέβασαν κάποιες ε, ε, τροπολογίες και είπαμε ότι αυτέ θα συγκεντρώσουν ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με την έκθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά τρίτον είπε ο συγκριτής ότι θέλουμε να ε, μάτιωθούν όλες αυτές ε, ε, οι περικοπές σε σχέση με το πρόγραμμα για το 2020 και όσον αφορά την ευρωδιευκόλυνση το Connecting Euro Facility και είπαμε στο 1 ε είπαμε να μάτιωθούν όλες οι περικοπές του Συμβουλίου και να χρησιμοποιήσουμε ό,τι περιθώριο και υπάρχει τόσο ώστε να ρίξουμε τις ΜΜΕ και αυτό επίσης να βοηθά ε, όπως βοηθούν και κάποια μέτρα, ε, ε, έρευνα όπως το πρόγραμμα Μαρία Κιουρί, η έρευνα, το Ερευνητικό Συμβούλιο, το Έρασμος, το κόσμε, όπως είπαμε έρευνα και μη μία θεωρούμε ότι ό,τι υπάρχει τώρα ως ε, αποθεματικό να χρησιμοποιηθεί για αυτό τον σκοπό. Μέτρα δημιουργίας απασχόλησης. Πρωτοβουλία για ε, απασχόληση των νέων έχουμε μια τροπολογία και λέμε ότι η χρηματοδότηση για αυτή την πρωτοβουλία για το 2017 θα πρέπει να μείνει στα ίδια επίπεδα όπως ε, και κατά την περίοδο 2014-2015 αρχή του ισχύοντος ε, MFF. Και ακούσαμε χθε από τον κύριο Γιούγκερ ότι αυτή η πρωτοβουλία βοηθά τους νέου. Και έτσι μπορούν να βρουν κάποια δουλειά, μπορούν να κάνουν κάποιο είδου ε, stage, stage, δοκιμαστική περίοδο, δηλαδή μαθητεία και άπαξ και ε, δεν έχουμε κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την κάλυψη κάποιων προβλημάτων για την πρωτοβουλία γιατί η χρηματοδότηση και η πρικοδότηση να μην αξιοποιηθεί. Οπότε αυτό το ένα δις που προτείνει η Επιτροπή για το υπόλοιπο MFF θεωρούμε ότι είναι δεκάδες. Και γι' αυτό η δική μας αφετηρία είναι ακριβώς ό,τι περιέχει η έκθεση olbricht Τομά. Οπότε, το Ευρωπαϊκό Λεγό Κόμμα έχει κατεβάσει κάποια τροπολογία και προτείνουμε αύξηση κατά 4 εκατομμύρια για το Ταμείο με α, τους, ε, τους μη προνομίχους της Ευρώπης οπότε είπαμε ότι δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθούν, να το ξεχάσουμε. Στη ε, τίτλο 2 έχουμε επίσης μία τροπολογία που αναφέρει και ο εισηγητής 500 εκατομμύρια ευρώ υπέρ των γαλακτοπαραγωγών. Αυτοί που έχουν χτυπηθεί από την κρίση στον κλάδο τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει ε, την σχετική τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού, αλλά είναι σημαντικό να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς τους γαλακτοπαραγωγούς. Δεν πρόκειται περί συμβολικής χειρονομίας. Είναι πολύ σημαντική πολιτική πράξη. Οπότε και εμείς προσδοκούμε ότι αυτή η οικονομική στήριξη των όσων ευθύγησαν από την κρίση θα είναι θέση του Κοινοβουλίου όπως και η δεύτερη τροπολογία την οποία προτείνουμε όπου λέμε για 100 εκατομμύρια για τους γαλακτοπαραγούς που έχουν χτυπηθεί από το ρωσικό εμπάργκο. Επίσης ε, έχουμε ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα στο κεφάλαιο τρία που είναι χαμηλές οροφές, οπότε θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερο προσωπικό η Europol γιατί θέλουμε να βροντίσουμε την ε, ασφάλεια της Ευρώπης αυτό θέλει ο κόσμος στο τρίτο κεφάλαιο επίσης έχουμε πει για κάποιες μικρές αυξήσεις για την πολιτική γειτονία προς Ανατολάς και σε σχέση με την Μεσόγειο οπότε θέλουμε και οι δύο αυτές πολιτικές ε, γειτονίασεις να θεωρηθούν προτεραιότητες του Κοινοβουλίου γιατί θα πρέπει να ξέρουμε σε τι κόσμο ζούμε, τι γείτονε έχουμε. Έχουμε την Ρωσία, όλο ένα πιο επιθετική, έχουμε την Ουκρανία που έχει τόσο αποσταθεροποιηθεί, έχουμε την Τουρκία που είδαμε τους τελευταίους μήνες πόσο λίγο μπορούμε να την εμπιστευόμαστε, έχουμε τη Μέση Ανατολή, έχουμε επίσης και την ε, Βόρεια Αφρική. Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς θα πρέπει να φροντίσουμε τα της γειτονιάς μας και προς Ανατολάς και προς Νότον. Οπότε κατεβάσαμε αυτή την τροπολογία για να υπάρξει η μακροοικονομική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Και θεωρούμε ότι ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει η περικοπή 2016-2017 από την Κομισιόν από 80 σε 30 εκατομμύρια. Θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη αυτή η περικοπή, οπότε και εμείς λέμε να μην πάει από 30 σε 80, αλλά να πάει από 30 σε 35. Κάτι το οποίο συνάδει και με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ίντα, που είναι η κυρίως αρμόδια για το θέμα. Παρακαλώ. Σας ανέφερα τις βασικές ε, γραμμές, της θέση της ομάδας μας και βασικά συμφωνώ με τον εισηγητή. Υπάρχουν όμως δύο σημεία. Επ' αυτών προς το παρόν δεν συμφωνούμε με τον εισηγητή. Είναι σημαντικά σημεία για το ΕΛΚ. Σας εξηγώ. Πρώτα πρώτα. Στο αποθυματικό χρήματα για το ΕΦΣΙ. Ξεκάθαρα σας λέω ότι δεν θα συμφωνήσει με αυτό η πολιτική μας ομάδα. Είναι κόκκινη γραμμή για μας. Και εξηγούμε. Το ΕΦΣΙ είναι κάτι νέο. Διανύει την πρώτη του χρονιά. Ακούσαμε μέχρι τώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι αξιολογήσει. Δεν έχουμε άλλε αξιολογήσει. δεν έχουμε κάτι άλλο το επίσημο το οποίο να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα. Μπορεί να βελτιωθεί, μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσει, προσθετικότητα, να έχει ίσως ε, κανόνε παιχνιδιού για όλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μα αυτό θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποιε ε, προτάσεις της που αφορούν ακριβώς την προσθετικότητα Και ας πούμε, αν κρυθεί έτσι, δεν θα χρηματοδοτείται ένα αυτοκινητόδρομο στην Γερμανία και θα πηγαίνουν τα λεφτά εκεί που υπάρχει ανάγκη. Σε κάποιε γωνίες δηλαδή, τη Ευρώπη που χρειάζονται πραγματικά οι πόροι. Τώρα δηλαδή υπήρχε αυτό το θέμα, αυτή η διαφορά μεταξύ παλιών και νέων κρατών μελών όσον αφορά κάποια χρηματοδοτικά μέσα, κάποιες εταιρικές σχέσεις ή κάποιες επενδυτικές τράπεζες εμπορικέ τέλο πάντων και αυτά όλα τα έχουν υπόψη μα. Και διαπιστώνουμε ότι η Τράπεζα Επενδύσεων και η Επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν τόσο στον ίσιο όριο ανταγωνισμό και αυτέ οι διαφορέ, οι ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών να λιανθούν. Και για τι ΜΜΕ θέλουμε να βοηθήσουμε να υπάρχει απασχόληση, εκεί πάει καλά. Και έχουμε τι προσαρμογέ που επιφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που που ε, είναι κάτι το λογικό, αλλά είπαμε να στείλουμε το σωστό μήνυμα προς ΜΜΕ, προς θετικό τομέα. Να υποστηριχθούν οι εταιρείε και κυρίως οι ΜΜΕ. Το σχετική θηρίδα τα πάει πάρα πολύ καλά. Προσοχή μην είμαστε αντιπαραγωγικοί όμως είπαμε, αυτός είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό και λέμε να μην πάνε πόροι του εύσης στο αποθεματικό. Τελευταίο. Άμυνα. ...της ε, προπασχεδευτής δράσης για την άμυνα. Άρα επ' αυτού συμφωνούμε τον εισηγητή. Όμως, μην ξεχνάμε ότι 50% από αυτά τα χρήματα που θα πάνε σε αυτές τις δράσεις θα πρέπει να πάνε στις νέες πρωτοσκευαστικές δράσεις να αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε εάν ε, για την άμυνα αυτές οι πρωτοσκευαστικές δράσεις θα οδηγήσουν σε καλύτερη έρευνα, σε καλύτερη καινοτομία άμυνα και έτσι θα αναβαθμίσουμε τις ε, αμυντικές μας ε, δυνατότητες. Για μας αυτό είναι προτεραιότητα και νομίζουμε πρόεδρε ότι έτσι θα πρέπει να έχουν τα πράγματα και εδώ θα βάλω τελεία πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο συνοπτικός, διότι πρέπει να τη δέκα να έχουμε κλείσει. Ευχαριστώ. Αληθεύει ότι για τα άλλα τμήματα μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε τις προτάσεις ε, για το προϋπολογισμό συμφωνούμε φυσικά με τις δεσμεύσεις ε, της πενταετής για τη μείωση κατά 60 θέσεις ε, Επίσης, ε, συμφωνούμε για τις θέσεις ε, που δεν επιστράφηκαν στην Επιτροπή των Περιφερειών, το αντίθετο, και υπέρ των 35 θέσεων για τα θέματα ασφαλείας και για το αμφιλεγόμενο ζήτημα για τις 76 πολιτικές, νέες πολιτικές θέσεις, γιατί δεν είναι μόνο μια διοίκηση, το Κοινοβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο, κατεξοχήν κιόλας. Οπότε νομίζω θα πρέπει να καλύψουμε αυτό το κενό. Για τα υπόλοιπα τιμήματα, Όντω. για το δικαστήριο, αλλά για το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να αποκαταστήσουμε τις γραμμές ε, ε, και το ίδιο για ε, τον διαμεσολαβητή και για τον επόπτη προσωπικών δεδομένων. Για το δικαστήριο πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις 12 θέσεις για τους δικαστές. Έτσι, Κάθε χώρα θα έχει το δικό της δικαστή. Για την ΟΚΕ και για την Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να επανεντάξουμε όντω τι θέσει που δεν επιστρέφηκαν στο Κοινοβούλιο 12 και 8 αντίστοιχα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό όπως και αν το δει κανεί. Επίσης, για τους μισθούς η μείωση είναι κάτι ε, που είναι ένα έτοιμο που θα πρέπει να ικανοποιήσουμε γιατί το περιμένει το προσωπικό. Και ανάμεσα στους αποσπασμένους για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και τους ε, υπαλλήλου. πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Οπότε ναι για τη δημιουργία νέων, 16 νέων θέσεων. Αυτή η μονάδα για την στρατηγική επικοινωνία μου φαίνεται πολύ λογικό, ε, πολύ λογικό βήμα για να κρατήσει αφήνει για διάφορα ζητήματα. Ξαναλέω, για τις 76 πολιτικές θέσεις επιμένουμε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι μάλλον πολιτικό παρά διοικητικό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, Κόλμελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας... Ε, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έκαναν τόσο μεγάλη δουλειά ε, προπαρασκευαστικά και κυρίως τον κύριο Γκάιερ θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί πραγματικά όλα όσα μας ανέφερε ήταν πολύ εμπεριστατωμένα. Και συμφωνώ απόλυτα στην, με την ανάλυση σας και με την αξιολόγησή σας ό,τι αφορά το ΕΦΣΥ που κι εσείς κύριε Γκάιερ πιστεύετε ότι υπάρχει ε, κίνδυνος να χάσουμε μεγάλο κομμάτι της διαφάνειας. Συμφωνώ δε και με το ότι δεν θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με κάποιες γενικές αφηρημένες περιγραφές. Και επιτρέψτε μου λοιπόν στο σημείο αυτό να κάνω και ένα μικρό παλληλισμό. Εντάξει, δεν είναι ταυτόσιμος ασφαλώς, αλλά είναι ένας καλός παραλληλισμός. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κατά την ίδρυσή της, τι είχε γίνει. Ήταν σαφής ε, σχετικά οι κανόνες λειτουργίας της. Αλλά εν τω μεταξύ υπάρχουν ε, νέα μέσα χρηματοδότησης, ε, μη συμβατικές τοποθετήσεις και ισορροπίες. Φοβάμαι λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά ένα μέσο όπως το ΕΦΣΥ αν λάβει τέτοιε ε, διαστάσει, ε, θα υπάρχουν πολλά ταμεία, όπω για παράδειγμα το Ταμείο για την Αφρική και πολλά άλλα, όπου θα έχουμε κάποιε εγγυήσει, αλλά όλα τα υπόλοιπα θα είναι εκτό του πεδίου αρμοδιοτήτων μα και εμεί απλά θα είμαστε τελευταίοι και καθαϊδρωμένοι. Άρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να αγωνιστούμε για να έχουμε δικαίωμα υποπτία επί του ταμείου αυτού. Και κατά τα άλλα θα πρέπει να σας πω και να μιλήσω για δύο α, τροπολογίες του ECR. Η μία έχει να κάνει με το ότι θεωρούμε ότι και σε θέματα πολιτικής συνοχής δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε πάνω στον την πορεία την οποία έχουμε ακολουθήσει έως τώρα και άρα θέλουμε να έχουμε καταθέσει τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. για να υπάρχει κάποια μεταφορά, αν θέλετε, των πόρων προς τις λιγότερο αναπτυσσόμενες περιοχές που έχουν πιο πολύ ανάγκη τους πόρους αυτούς. Και ύστερα τους πόρους ε, που προβλέπονται για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ένα τμήμα των πόρων αυτών να πάει στο αποθεματικό. Γιατί ξέρουμε ότι στην παρούσα φάση αυτή η συμφωνία δεν έχει υλοποιηθεί και υπάρχει και η ανησυχία, ο φόβος ότι δεν θα υλοποιηθεί καν. Και άρα θεωρώ ότι πολιτικός πώ θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα. Ευχαριστώ κύριε Τεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγχαρητήρια στον κύριο Γκάιερ και στους συνεργάτες του. Είναι εξαιρετικά ποιοτικό το έγγραφο και ήταν και πολύ ε, λίγος ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για να διάφορους προβληματισμούς. Όταν αναλύω λοιπόν το κείμενο, κυρίως για την κατηγορία 1α, επειδή εμείς είχαμε καταθέσει πολλές τροπολογίες. Διαπιστώνω ότι εδώ πέρα ε, είναι οι σοσιαλιστές, έλκα, σοσιαλιστές, έλκα, σοσιαλιστές, έλκα, σοσιαλιστές, έλκα, σοσιαλιστές, έλκα, σοσιαλιστές, έλκα. είναι οι τροπολογίες που εγκρίθηκαν. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει. Τεχνικής φύσης είναι το πρόβλημα. Εμεί για όλες τις γραμμές καταθέσαμε τροπολογίε. Ήταν να κάνουν μόνοι τους το ΕΛ σοσιαλιστές στον προϋπολογισμό τότε. Μην ε, εκπλήσονται όμως αν κάποιοι άλλοι δεν τους υποστηρίζουν. Ε. Θέλω μια λογική εξήγηση, διότι όποιο και ένα τεχνικός λόγος δεν μου φαίνεται σωστό. Να πει ο εισηγητής ότι είναι συμβαστική τροπολογία και να αναφερθεί σε όλες τις τροπολογίες που μας οδήγησαν στη συμβαστική. Όμως, η πρωτοβουλία για τους νέους, πάλι τα ίδια. ΕΛΚ, ε, σοσιαλιστές, ε, για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ΕΛΚ, σοσιαλιστές. Οι άλλοι δεν έχουν καταθέσει τροπολογίες. Δεν θέλω, δεν πρόκειται τώρα για ε, ε, σταυροφορία. Αλλά Εάν δεν υπάρχει αντικειμενικό τεχνικό λόγο δεν μπορώ να το δεχτώ. Ήθελα να το πω εξ αρχή και να είμαι σαφή. Δεύτερον, ποτέ δεν ήμουν υπέρ, ακόμη και όταν ήμουν εισηγητή, ποτέ δεν ήμουν υπέρ τη δημιουργία 76 νέων θέσεων για τι πολιτικέ ομάδε. Θα αντιταχθούμε. Με τη χτενισινή συζήτηση είδα ότι υπάρχουν δύο σχολές. Αυτή που είναι κάθετα εναντίον και άλλοι που λένε, α, θέλετε 76, τότε θέλουμε αντιστάθμιση. Αυτές οι δύο θέσεις είπαμε, αυτές οι δύο σχολές. Θα είναι κόκκινη γραμμή για την ομάδα μας. Αυτές οι προκατακτικές παρατηρήσεις και τώρα στην ουσία. Συμφωνώ με τον προσανατολισμό του κ. Γκάιερ. Να αποκατασταθούν όλες οι γραμμές που έκοψε το Συμβούλιο. Δεύτερον, αν κατάλαβα καλά, συμφωνώ με τη στρατηγική του Δηλαδή για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλία για τους νέους και για την αποκατάσταση των πιστώσεων ορίζοντας 2020 και ΣΕΦ από, τις, από τα επιπρόσθετα κονδύλια που πήραμε από την ενδιάμεση αναθεώρηση. Αν ε, δεν κατάλαβα καλά, παρακαλώ διορθώστε με. Αν κατάλαβα καλά, συμφωνώ. Για τις ε, πληρωμές, να το συζητήσουμε, να έχουμε πιστώσεις πληρωμών που ε, ε, ε, αντιστοιχούν στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Δεν υπάρχει πάντα τεχνική αιτιολόγηση, αλλά μπορούμε να το καταλάβουμε σε πλαίσια μια συνολική στρατηγικής με απότερο στόχο να αυξηθεί το επίπεδο των πληρωμών, διότι είχαν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. συγγνώμη, προσπαθώ να είμαι σύντομος, αλλά είναι πολλά. Έχουμε ενδιασμούς. Όχι για το, τα να μπουν τα κονδύλια του ΕΦΣΙ στο αποθεματικό, αλλά διότι δεν καταλαβαίνω. Βάσει ποια, ποιων αντικειμενικών ε, κριτηρίων θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Μιλάτε για την προστατικότητα και για την εξορροπημένη κατανομή. Καμία σχέση. Είναι θέμα πολιτικής ερμηνείας. Δεν πιστεύω στην αντικειμενική στην αντικειμενικότητα της διαδικασίας που μας ε, επέτρεπε να άρουμε την επιφύλαξη για το αποθεματικό. Χρειάζεται εναλλακτική λύση επίσης για τα 25 εκατομμύρια που ζητάει η Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να θέσω κι άλλο ένα ερώτημα. Δεν είδα σχεδόν πουθενά εκείνο είναι θέμα αρχής και πάλι. Υπάρχει ίσως λογική εξήγηση ο, η ομάδα μας κατέστησε πολλές τροπολογίες, κυρίως ο κύριος Τόρβαλς ζήτησε αύξηση των πιστώσεων τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο να υπάρχει, ε, ε να προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα μετά την COP21. Δεν είδα τίποτα. Είναι μάλλον κάτι αστείες παραχωρήσεις που γίνονται μάλλον για τους πράσινους. Στο heading 2, 17 εκατομμύρια. Ψίχουλα. Ένα β. Θέλω να εξηγήσω για ποιο λόγο ζητήσαμε προς το κονδύλι για την πρωτοβουλία. Θεωρούσαμε ότι υπάρχει αντικειμενικό λόγο να μπει στο αποθεματικό. Αφού πριν το τέλο του τρέχοντο θα κάνει την αξιολόγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε είναι αποτελεσματικό αυτό ο μηχανισμό, χρειάζεται αναπροσαρμογή. Αυτό είναι όμω λόγο για τον οποίο ζητούμε το ποσό αυτό να μπει στο αποθεματικό. Αλλιώ Συμφωνώ με τον εισηγητή. Τμήμα 2. Συμφωνώ με τον κύριο Κρεσά από πλευράς ΕΛΚ. Θέλουμε να μπουν τα κονδύλια στη γραμμή. Αν περιμένουμε το διαστηματικό προϋπολογισμό, μετά τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τμήμα 3. Πρόεδρε, Ε, Μα αρέσουν οι ιδέε σα, αλλά έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ε, ε, Eurojust, ωραία. Το ψήφισε η Λίμπε. Τα 5 εκατομμύρια εγώ δεν τα είδα στην ψηφοφορία στη Λίμπε. Από πού μπορεί λοιπόν αυτό το αίτημα, αφού στην ψηφοφορία στη Λίμπε δεν τα είδα αυτά τα εκατομμύρια. Να ε, επισημάνω κάτι που είναι περίεργο. Ε, στο τμήμα 3 έχουμε τα μεταναστευτικά προβλήματα, τα προβλήματα ασφάλειας και πρέπει να κινητοποιηθούμε, να είμαστε σε γρήγορος και να έχουμε επιπρόσθετα μέσα. Όμως, εάν ε, διαβάσουμε τις προτάσεις που θα καταλογιστούν στο Κοινοβούλιο για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, Europol, Eurojust και ούτω καθεξής, θα ζητήσει 11 επιπρόσθετα εκατομμύρια το Κοινοβούλιο. Αντίθετα, για την ηθαγένεια και τον πολιτισμό παίρνω όλα τα Δεν λέω ότι με κατά, απλώς ρωτάω. Ζητάει 47 εκατομμύρια το Κοινοβούλιο και ρωτώ. Από πολιτικής ε, σκοπιάς ε, ε, έχει κάποιο νόημα, δηλαδή το Κοινοβούλιο ζητά 11 επιπρόσθετα εκατομμύρια για τη μετανάστευση και την ασφάλεια και 47 εκατομμύρια για τον πολιτισμό. Νομίζω καλό είναι να ρωτηθούμε. Τμήμα 4. Έχω τεχνικού χαρακτήρα παρατηρήσει αλλά δεν είναι η σωστή στιγμή του σωστό Τμήμα 5. Σας είπα και πριν, θα, έχετε, θα σας δημιουργήσουμε δυσκολίες με αυτές τις θέσεις ε, που θέλετε. 114 σοφέρ, 76 πολιτικές θέσεις, 35 για την ασφάλεια συμφωνούμε. 225 νέες θέσεις, ενώ από όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα ζητάμε ε, να κάνουμε περικοπές προσωπικού 5%. Εγώ δεν μπορώ να υπομιστώ την πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Ευχαριστώ. Μεριέντα. Δεν θα ακρηγορήσω. Ευχαριστούμε κύριε Γκάιερ. Μας δώσατε μια εικόνα του πώς έχουν τα πράγματα και θα ήθελα να προσέξετε το ένα α και τα 2 κονδύλια σε αυτό το τομέα τμήμα. Λέμε για τις περιοχές που πρόκειται να φυγούν από το Brexit. Ξέρω ότι έχετε βαρεθεί να μην ακούτε, αλλά θα γίνει κάτι τέτοιο, θα υπάρξει κρίση. Σε Σκοτία σε Βόρεια Ιρλανδία, σε αυτούς που θα είναι μέλος, μέρος συγγνώμη, του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις περιοχές στην τύχη τους. Θα πρέπει αυτά τα δύο κονδύλια να αυξηθούν. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δείξει στον κόσμο ότι δείχνει την αλληλεγγύη του, την αλληλεγγύη γιατί η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη Λέμε για στρατιωτικοποίηση και ευρωπαϊκό στρατό. Μα για να γυρίσουμε στο α, στην αφετηρία μας. Γιατί φτιάξαμε την Ευρώπη. Να δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση και ότι το Κοινοβούλιο θέλει την ειρήνη. Να μην ξεχνούμε ότι το Κοινοβούλιο είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Και ε, αυτή η ειρηνευτική διαδικασία πρόκειται να υπονομευθεί από τον Brexit. Άρα χρειάζεται και για τη Σκοτία και για την Βορειοελλανδία ενίσχυση. Αυτό λέμε κι εμείς. Να μην τους αφήσουμε στην τύχη τους, γιατί η Αγγλία αυτό θα κάνει. Θα τους αφήσει στην τύχη τους. Είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται σε κάποιες δαπάνες όπως το πρώτο τμήμα. Εμεί θέλουμε να υπάρχουν ε, τα προγράμματα για την απασχόληση, θα πρέπει να επανέλθει σε κάποιες περιπτώσεις ε, ό,τι προτείνει η Επιτροπή, αλλού θα πρέπει να αυξηθούν αυτά που προτείνει η Επιτροπή, θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας για την απασχόληση που είναι προτεραιότητα. Επίσης θα πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Όχι, δεν θέλουμε τα χρήματα για το ΕΦΣΙ να πάνε στο αποθεματικό. Και θα πρέπει να αυξηθεί η οικονομική στήριξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Ε, κατάρτιση, έρασμος, όλα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν Συμφωνώ με τον κύριο Γκάιρ που είπε για ενίσχυση προς τη δική μου χώρα και για τα πολιτιστικά να δημιουργήσουμε μέσω του πολιτισμού απασχόληση. Για κάθε οικονομία βέβαια και για τη δική μας είναι πολύ σημαντική τομής η αλία και ο λακτομικός τομέας οπότε και αυτούς θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Ε, να καλύψουμε πρόσφυγες και μετανάστες με τα σχετικά προγράμματα και με κάθε σεβασμό όλα αυτά τα οποία προτείνονται για την ασφάλεια μήπως θα έπρεπε αυτά να πάνε κάπου αλλού που να είναι κάτι πιο θετικό κάτι που να βοηθά ε, στους σκοπούς και στους στόχους για τους οποίους φτιάχτηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και δίνω το λόγο στον κύριο Μαραγκάλη. Πρώτα πρώτα. Α, έφυγε ο κύριος Γκάιρο όμως. Τέλος πάντων, εγώ τον ευχαριστώ ούτως ή άλλως για την εισήγησή του και για τη δουλειά του. Επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες, νομίζω θα τα πούμε και θα τα βρούμε και θα έχουμε σύγκληση θέσεων που φαίνονται ότι αποκλίνουν. Δύο πολύ βασικά. Πρώτα πρώτα ο συμβιβασμός, η δέσμευση για τις τροπολογίες μας πέρασαν και εγκρίθηκαν από κάποιες επιτροπές. Άρα αυτές οι τροπολογίες θα προχωρήσουν. Επίσης ε, συμφωνούμε με την θέση Γκάιερ που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των κονδυλίων που προτείνονται και κόντρα στις περικοπές του Συμβουλίου. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτό, κάτι άλλο έχω να προσθέσω. Να συνεχίσουμε να έχουμε υπόψη μας την δέσμευση του Ιουλίου της Επιτροπής μας. Αυτό το οποίο μπήκε στις κατευθυντήρες γραμμές για την χρήση 2017 και σε σχέση με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, το MFF. Θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε και για την συνέπεια της θέσης μας και αυτό ότι καταδώσουμε κάποιες τροπολογίες επίσης για το έρασμος συμφωνούμε με τον κύριο Γκάγερ αλλά επίσης συμφωνούμε για το ΕΦΣΕ θα τον υποστηρίξουμε 100%. Επίσης, ανησυχούμε σε σχέση με το εύση, με αυτά που έχουν πει και θα πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία προτείνει ο συγητής. Να υπάρξει πάντως τελικά ένα πρόγραμμα επενδύσεων πραγματικό γιατί το έψη ακόμα δεν είναι τέτοιο. Θα πρέπει να δεχθούμε ή να μην δεχθούμε τις θέσεις της κυρίας Γεωργίβα για το MFF. Να λάβουμε υπόψη ότι ταυτόχρονα έχουμε τις εξελίξεις στους ιδίους πόρους. Αυτό έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες ως εξέλιξη. Και επίσης έχουμε το θέμα των δημιουργικών επιδόσεων της ευρωζώνης Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ίσως δεν έχει ληφθεί ακόμη υπόψη, αλλά σύντομα θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, συμφωνώ με τα όσα λέει ο κύριος Γκάιερ για την προπαρασκευαστική δράση για την άμυνα νέος στόχος. Ε, κατά κάποιο τρόπο μπαίνει αυτός ο στόχος στο παιχνίδι μέχρι τώρα από την πίσω πόρτα, την γερκό πόρτα, αλλά όχι, όχι. Να μπει από την κυρία είσοδο. Είναι δέσμευση των κρατών μελών. Θα πρέπει να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους που δεν το έκαναν στο παρελθόν. Οπότε γι' αυτό και νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλει ο εισηγητής και συμφωνούμε για αυτήν την προπαρασκευαστική δράση. Έχουμε 28 τροπολογίες. Μπορούν να χωριστούν σε 5 ομάδες. Πρώτη ομάδα. Έχουμε κάποιες τροπολογίες που κατέβηκαν γιατί θέλουμε ήδη μέσα στο 2017 να αναθεωρηθεί το MFF. Αυτό το οποίο είπαμε στην έκθεση του Ιουλίου. Αυτό συνεχίζουμε να πρεσβεύουμε. Επίσης, σημαντικές αυξήσεις, λέμε στην άλλη ομάδα τροπολογιών, αυτά το που είπαμε στο έγγραφο πλαίσιο, ε, European Initiative, Έρασμος, ε, Δημιουργική Ευρώπη, ε, Ευρωπαίος πολίτης με μετανάστευση κλπ. Οπότε και έχουμε τώρα 4 εκατομμύρια και κάτι. Και έχουμε επίσης και 700 και 710 χιλιάδες από την άλλη μεριά. Και όλα αυτά περιέχονται στην έκθεση Olbricht Toma. Να αρχίσει η αναθεώρηση του MFF το 2017. Ε, η αύξηση είναι 3% μόνο, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε και να υπάρξει επίση κάποιο περιθώριο ευελιξία. Ένα, ένα λεπτό, πρόεδρε, ένα λεπτό. Στην τρίτη ομάδα τροπολογιών μα. Εκεί θέλουμε το Horizon 2020 να αποκατασταθεί και το Connection Europe Facility να στα επίπεδα ε, στο 1.250 στα επίπεδα τα παλιά. Και επίσης και έχουμε και κάποια άλλα πράσινα ε, πράσινα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν Και στην ε, τελευταία, στη τελευταία ομάδα τροπολογιών έχουμε κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, Citizens Initiative, κάποιο αποθεματικό για τον κώδικα ε, διοντολογίας, ασφάλεια, μετανάστευση Frontex και αυτά. Και αυτά είναι σημαντικά, Πρόεδρε. Οπότε νομίζω ότι θα, δουλέψουμε καλά, γιατί έχουμε πάει μέχρι τώρα. Αναφέρει ο κύριος Ντεπρέ σε κάποιο έγγραφο του ΕΛΚ που είναι νομίζω αξιόλογο σαν ε, ε, αφετηρία. Συμφωνούμε. Ε, πρέπει να δούμε ξανά την παρουσίαση, αλλά νομίζω ότι τα ποσά θα πρέπει να τα δούμε και νομίζω ότι τελικά θα συμφωνήσουμε. Επόμενο, πάρα πολύ γρήγορα και σε, ευχαριστούμε και εμεί ευχαριστούμε τον εισηγητή. Η πρώτη μας γενικόλογη σκέψη για την προσέγγιση που ακολούθησε εκείνο. Το Συμβούλιο με αυτό το οποίο προτείνει καθόρισε κάποιες προτεραιότητες. Έστειλε ένα μήνυμα στο τι πιστεύει, που θεωρεί ότι πρέπει να μπει στον προπολογισμό και τι θεωρεί ότι δεν πρέπει να μπει. Αυξάνονται κάποια κονδύλια και θα πρέπει τα κράτη-μέλη όλα αυτά να τα υλοποιήσουν. Βέβαια έτσι ε, αλλάζεται τελείω η υπόθεση της Κομισιόν. Θέλει το Συμβούλιο της ε, περικοπές και δεν νομίζω ότι δίνει τώρα μια καλύτερη λύση από την Κομισιόν. Τώρα για κάποια συγκεκριμένα σημεία ε, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι θα υπάρξει αποκατάσταση κάποιων ε, ειδικών χρηματοδοτικών μέσων. Το είχαμε και εμείς ζητήσει αυτό, ε, αλλά μας προβληματίζει κάτι το οποίο ακούσαμε, δηλαδή το τι θα γίνει με το ΕΦΣΙ και επίσης αυτό το οποίο είπε χθε ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράταση ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείο για τις ε, επενδύσεις και επίσης το τι θα γίνει με το ΕΦΣΙ και τις τρίτες χώρες. Οπότε έχουμε κάποιους πόρους για τα σχετικά προγράμματα. Θεωρούμε όμως ότι έτσι θα δημιουργηθεί πίεση στις επόμενες χρήσεις, στους επόμενους προϋπολογισμούς. Αυτή είναι η γενική μας ε, σκέψη. Τελευταίο τώρα, ο, κάτι που θέλουμε να τονίσουμε αφορά την Τουρκία. Είναι γνωστό το τι συνέβη το καλοκαίρι. Βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση Ερντογάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα στην Τουρκία και να υπάρξει πλήρης και ρεαλιστική αναθεώρηση ε, των χρημάτων που έχουμε δεσμευτεί. Ε, αυτά τα οποία στέλνει η ΕΤΕ στην Τουρκία θα πρέπει επομένω να δούμε ότι μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα αποφασιστικό, ε, τίποτα ουσιαστικό, αλλά θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη τώρα όσον αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Βεβαίω και συμφωνούμε με αυτά που λέει ο εισηγητή όσον αφορά αυτές τις 76 θέσεις απασχόλησης για τις πολιτικές ομάδες. 2 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά θα δαπανηθούν ίσως ε, δεν είναι αύξηση προτεραιότητας για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Ακόμα εκκρεμούν πάντως άλλα θέματα για την εσωτερική υπηρεσία των σοφέρ και την πρόσληψη ως υπαλλήλων τούτων. Πρόκειται για κάποια ιδέα που βρίσκεται εν εξελίξη. Ίσως θα πρέπει και επ' αυτού να προβληματιστούμε γιατί είναι κάτι το απαραίτητο είναι το μοναδικό κονδύλιο το οποίο εκθετικά αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Ε, καλό σημάδι είναι αυτό. Όσον αφορά πάντως τις ε, περιφερειακές υπηρεσίες ίσως είναι το καλύτερο να γίνουν και εκεί περικοπές όπως προτείνεται. Ο ρόλος πολλών τέτοιων υπηρεσιών θα μπορούσε να υποκατασταθεί από γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν. Θα μπορούσαμε να είχαμε εκλογήκευση της κατάστασης με αυτές τις περιφερειακές υπηρεσίες. Ίσως αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να το κάνουμε. Και το ίδιο ισχύει ας πούμε όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, όσον αφορά την Επιτροπή τη, ε, την Περιφερειακή Επιτροπή και επίσης θα πρέπει να δούμε Ποιος ήταν ο μελλοντικός ρόλος αυτών των υπηρεσιών. Ίσως αυτό θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση του ρόλου τους και όχι η περικοπή. Και το θα πρέπει επίσης να δούμε και τι θα γίνει και με την, με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Euh, Παρακαλώ να είστε σύντομοι, ναι, θα είμαι γιατί έχει περάσει η ώρα. Ε, υποστηρίζω τον εισηγητή, έχει κάνει σκληρή δουλειά, κυρίως ε, για το ΕΦΣΥ και την αποκατάσταση των γραμμών. Και το θέμα της λογοδοσίας ε, σε όποιο τομέα μπορούμε και την προπαρασκευαστική δράση τα υποστηρίζουμε. Να ξέρουμε από πού έρχονται τα κονδύλια και ποιο είναι το κίνητρο. Το ε, θέμα είναι η υποστήριξη για ε, τα μέτρα για το προσφυγικό και η υποδοχή των πρόσφυγων. Ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου να κάνω και εγώ κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις. Εξαιρετική δουλειά έκανε ο Γενικός Ανσηγητής και Συγητής για τα επιμέρους τμήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και νόμιζα ότι πρέπει να κλείσουμε στι 10.30, και αλλιώ θα είχα ζητήσει και εγώ το λόγο. και προφανώ ε, οι σοσιαλιστέ συμφωνούν ιδιαίτερω με τον κύριο Γκάιρ. Και νομίζω ότι σωστό θα ήταν να υπογραμμίσουμε κάποια στοιχεία εδώ πέρα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην, ε, στο τρίτο τμήμα. Γιατί εδώ έγιναν πολλές περικοπές και από πλευρά του, της Επιτροπής και από πλευράς του Συμβουλίου. Και σε ό,τι φορά το 4 το τέταρτο τμήμα νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες. Δεν θέλω να επεκταθώ τώρα σε ό,τι αφορά το πακέτο για την άμυνα. Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις, νομίζω ότι έχουμε μια καλή ευκαιρία να σκεφτούμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις μετά την αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και της διαθεσμικής συμφωνίας. Γιατί ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο προπολογισμό σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο τμήμα είναι ότι αφαιρούνται χρήματα από τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε στην Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει διστάθμιση με άλλες κατηγορίες και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια πρόταση παρόμοια. Αυτή είναι πιο μικρό επίπεδο, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Ο κύριος Φερνάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες στο σημείο αυτό, αλλά δεν ε, αισθάνομαι πραγματικά άνετα σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρίαση και δεν έχουμε λάβει κανένα έγγραφο. Ε, Ενδεχομένω, καλό να είναι το έγγραφο του κ. Γκάιρ, δεν λέω, αλλά δεν το έχουμε λάβει, δεν έχουμε ενημερωθεί και όλη αυτή η συζήτηση για τον προπολογισμό του 2017 θεωρώ ότι θα πρέπει να, να διεξαγάγεται υπό το φως των όσων διαπιστώσαμε στα πλαίσια του πολιτισμού συνομικού πλαισίου, τα αυτά που είδαμε χθε. Και εδώ λοιπόν κάποια γεγονότα με ανησυχούν ιδιαίτερω. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια αναδιανομή των πόρων. Σίγουρα υπάρχει αναδιανομή κάποιες από τις ε, δεσμεύσεις πληρωμών θα ε, αυξηθούν, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη συνοχή. Αλλά θα θέλαμε να δούμε ποιο σχέδιο υπάρχει σε ό,τι αφορά την περίοδο μέχρι το 2020 και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, ζητήσω την άλλη εβδομάδα που θα γίνει πάλι συνάντηση να λεφτεί υπόψη και, η μετα... και η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτές οι δύο συζητήσει θα πρέπει να συνάδουν. Ευχαριστώ πολύ και Φερνάντες. Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που υπάρχουν. Σίγουρα θέλει να λάβει υπόψη τις επιθυμίες όλων των πολιτικών ομάδων και έχουμε χρόνο ακόμη στη διαθέσή μας. Παρατηρήσεις. Αποθεματικό για το ΕΦΣΥ. Κάκι στο μήνυμα για τους επενδυτές. Οι συνάδελφοι ανέφεραν τους λόγους. Σύμφωνο με το Ζίγκφριντ μου αρέσαν το σκιώδι μας. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολιτικές ε, θέσεις. Κάποια στιγμή με την αναθεώρηση του πολιετούς, ε, το προϋπολογισμό 16 και 17, όλα αυτά θα συνδεθούν. Διότι η αναθεώρηση του πολιετούς θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό 16. και με τη στρατηγική μας, ε, δηλαδή να μην έχουμε τροπολογίες μας ε, συνάδουν με τη, τον προσανατολισμό μας για την αναθεώρηση του πολιετούς ε, και ακολουθούν και τις συστάσεις του εισηγητή. Ε, αυτή την προσέγγιση πρέπει να ακολουθήσουμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Ποια θα είναι η στρατηγική μα για να υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα τρία στοιχεία. Γιατί κάποια στιγμή θα κληθούμε να αποφασίσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάνδη. Δεν ζητάει κάποιο άλλο το λόγο. Χαιρετίζουμε τη δουλειά του εισηγητή. φόρο τιμή στον κύριο Γκάιερ. Θα περάσουμε τώρα στις πληροφορίες και τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και ε, είναι πολύ σημαντικό για μένα ε, να είναι σαφέστατο και εύληπτο το μήνυμά μας ε, και για τους πολίτες. Στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο θα έχουμε πειθό εάν Είμαστε συνεπείς και έχουμε ε, σαφείς προτεραιότητες. Θα αφήσουμε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και να ασχοληθούμε με ε, τις προτεραιότητες, τις πραγματικές προτεραιότητες. Και βασίζομαι στον συγητή και στους σκιώδες. Δεν πρέπει να είναι υπερβολικά πολλές οι προτεραιότητες για την ε, δράση κατά προτεραιότητα. Συμφωνώ με αυτούς που είπαν. Εντάξει, υπάρχουν ενδιασμοί και το σημειώνω. Ε, με αυτούς που είπαν ότι θα πρέπει η δράση να εκπέσει ε, του κονδυλίου για τα πολιτικά προγράμματα και τις ε, δράσεις προτεραιότητας. Γιατί μόνο έτσι θα πείσουμε το Συμβούλιο να κάνει μια κίνηση προς την κατεύθυνσή μας. Είμαι προβουλευτής όπως και εσείς και άρα επιτόπου εγώ θα κληθώ να εξηγήσω στους ψηφοφόρους μου τι ψήφισα εδώ. Προ το παρόν δεν έχω κανένα επιχείρημα για να αιτιολογήσω τη δημιουργία 76 νέων θέσεων για τις πολιτικές ομάδες. Οπότε δεν θα σας ξαφνιάζει να καταψηφίσω τι τροπολογίε. Είναι η προσωπική μου θέση. Είναι θέμα συνείδηση. θέλω να, έχω, να μπορώ να εξηγήσω στου ψηφοφόρου τι κάνουμε εδώ. Όταν όλοι μιλάμε για έλεγχο των δημοσίων δαπανών, α μην υποκύψουμε στο πειρασμό και την ψευδέστηση ότι κανείς δεν θα ασχοληθεί με αυτά που κάνουμε εδώ, γιατί θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά στο μέλλον. Ο εισηγητής για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Das würde jetzt das Zeitbudget... Νομίζω ότι αν ε, απαντήσω λεπτομερώς ε, στις ασχολητές των συναδέλφων, ε, δεν θα είχαμε χρόνο στη διάθεσή μας να τα πούμε όλα αυτά. σημείωσα πολλά από αυτά που σχολίασαν οι συνάδελφοι και στα πλαίσια των συντονιστών έχουν ζητηθεί πολλά τέτοια θέματα και έχει ε, δίκιο ο πρόεδρος Αρτουή με το έγγραφο αυτό και είναι αυτό έγγραφο εργασίας ε, Βρισκόμαστε στην αρχή μια διαδικασία. Ακούσαμε και αυτά που ακούσαμε χθε. Ε, προετοιμάζουμε και τις ε, επεξεργασίες, την επεξεργασία τον Οκτώβριο και σκοπός μου είναι να πετύχουμε μια στεναρή πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Γι' αυτό λοιπόν επιδεικνύω πνεύμα συμβαστικό. Το διαπιστώνετε αυτό, άλλωστε. Προκειμένου η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Αυτή την προσέγγιση λοιπόν θα ακολουθήσω και με τις ε, ομάδες, τις πολιτικές και είμαι αρκετά αισιόδοξη ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία όπως άλλωστε έχει συμβεί και στο παρελθόν. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη κύριε Γενική και εισηγητά. Μάλιστα. Και εσείς λοιπόν κύριε Τάραντ την ίδια άποψη έχετε. Μάλιστα πάρα πολύ ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις να πάρει συνεδρίασεις. Η επόμενη συνεδρίαση και η συνεδρίαση των συντονιστών και 26 Σεπτεμβρίου Δευτέρα έχουμε τους συντονιστές στις 28 ε, Σεπτεμβρίου από την 9 μέχρι το 10.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 5η 29 Σεπτεμβρίου 9 θα έχουμε την ψηφοφορία του προπολογισμού για το 2017. Στις 27 Σεπτεμβρίου που είχαμε μια συνεδρίαση έχει ακυρωθεί. Μάλιστα. Αυτά ε, κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτών για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών μετά.